Ε, διαπραγματεύσει για τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ. Δήλωση της Επιτροπής και θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Αλμούνια. Τον καλωσορίζω θερμά. Παρακαλώ. Κύριε Αλμούνια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Εξ ονόματος της Επιτροπής θα ήθελα να αναφέρω τους λόγους για επέκταση των εμπορικών μας σχέσεων με το Βιετνάμ, μια χώρα 90 εκατομμυρίων ανθρώπων, την τρίτη μεγαλύτερη της, Ενω... Ασίας, το 60 του ΑΣΕΑΝ. 60% είναι νέοι άνθρωποι μάλιστα. Εξάλλου το Βιετνάμ αναπτύσσεται πολύ θετικά, είναι πολύ επιτυχημένο και έχει μετατραπεί από μία από τις φτωχότερες χώρες σε μία χώρα μέσω εισοδήματος μέσα σε 25 χρόνια. Μπόρεσε να αναπτυχθεί σε ένα αριθμό 6% περίπου, μόλις κάτω από τα 6% ανάμεσα το 2008 και το 2012. Και πέρυσι για πρώτη φορά το Βιετνάμ ξεπέρασε την Ινδονησία όσον αφορά το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί τον τρίτο πιο σημαντικό ε, εταίρο μας μετά, ε, τέταρτο με συγχωρείτε, μετά από τη Σιγκαπούρη και την ε, την Μαλαισία και την Ταϊλάνδη. 90% δε της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης γεννάται εκτός της Ευρώπης στον τομέα της, νο, της Ασίας και του Ειρηνικού που υπάρχουν μεγαλύτερες, ε, πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου. Για μας στην Ένωση είναι λογικό να αυξήσουμε την εμπλοκή μας με τις ασιατικές οικονομίες ε, και με το Βιετνάμ. Παρά, ε, όχι μόνο τη, λόγω της δικής μας, του δικού μας ενδιαφέροντος, αλλά και με, ως τμήμα της στατηγικής ανάκαμψης. Υπάρχει ο απότερος στόχος της επίτευξης συμφωνίας με το σύνολο της περιοχής. Πέρα από τους δασμούς, η συμφωνία με το Βιετνάμ καλύπτει υπηρεσίε και, ε, και επενδύσει σε κρατικέ επιχειρήσει, δημόσιου διαγωνισμού και ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι διαπραγματεύσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί και θα υπάρξει σαφή σχέση ανάμεσα στις εμπορικές διατάξεις και τις πολιτικού τύπου διατάξεις για τη συμφωνία αυτή συνεργασίας που θα επιτρέψει στην Βιετνάμ να βασιστεί στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες προέβη όταν μπήκε στον ΠΟΕ για θέματα όπως η διαφάνεια, οι ε, διαβουλεύσεις ε, των εταίρων, έτσι όλα αυτά να συνδυαστούν με τις πραγματικές οικονομικές ανάγκες. Το Βιετνάμ προχωρά επίσης με ένα ευρύ επιλέγμα νέων συμφωνιών μέσω ευρύτερων διαπραγματεύσεων με το ΑΣΕΑΝ αλλά και μέσω της υπερειρηνικής ε, εταιρική σχέση. Ο, Επιτροπή, ο Επίτροπος Δεγκούχτ μετέβη στο Ανόη στις 17 Μαρτίου, όπου συναντήθηκε με τον Υπουργό Εμπορίου του Βιετνάμ, κάναν μια απογραφή της κατάστασης και ε, θέλουν να προχωρήσουν και να ολοκληρώσουν αυτές τις διαπραγματεύσεις ιδανικά πριν το πέρας του Οκτωβρίου ώστε οι επιχειρήσει ε, στην Ευρώπη και στο Βιετνάμ να μπορέσουν να αποκομίσουν τα ωφέλη και να δραστηριοποιηθεί η ανάπτυξη και στις δύο οικονομίες. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωκοινόβουλο για αυτό το ψήφισμα, το οποίο στέλνει σαφέ και συνεπέ μήνυμα στου εταίρους μας σε σχέση με αυτέ τι διαπραγματεύσει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πίτρο. Το λόγο έχει ο κύριος Κασπάρη, παρακαλώ. Αξιότιμη Πρόεδρε Κάρας, ε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Η συμμετοχή στο διεθνέ εμπόριο είναι πολύ σημαντική όταν πρόκειται για τη δημιουργία απασχόληση και ανάπτυξη. Και αυτό κατεξοχήν φαίνεται στι χώρε ΑΣΕΑΝ, τη νοτιο Ανατολική Ασία. Τι τελευταίε δεκαετίες άνοιξαν το εμπόριό του, συμμετέχουν στην παγκοσμιοποίηση και αυτό είναι ένα από του λόγου για του οποίου η οικονομική ανάπτυξη σε αυτή την περιφέρεια του κόσμου είναι τόσο ισχυρή. Εδώ και λίγα χρόνια έχουμε αυτέ τι διαπραγματεύσει με το Βιετνάμ και τότε η διαπραγματευτική εντολή ε, ήταν πάρα πολύ εντατική, συμπεριλήφθηκε η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού και με το σημερινό μα ψήφισμα φιλοδοξούμε μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει να θέσουμε προτεραιότητε που θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη σημερινή συζήτηση θέλουμε να δείξουμε και δημόσια ότι οι διαπραγματεύσει αυτέ, όπω και οι υπόλοιπε εξωτερικού εμπορίου γίνονται με όσο γίνεται πιο διαφανή τρόπο. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα επί της ουσίας είναι το εξής. Θα πρέπει αφενός να εξασφαλίσουμε ότι μέσω μακροπρόθεσμα το Βιετνάμ θα πρέπει ε, να έρθει κοντά μας είναι ακόμα πολύ αναπτυσσόμενη χώρα και με εντατικούς ρυθμούς αλλά ταυτόχρονα όλες οι εξαιρέσεις που προβλέπονται ε, και μεταβατικές περίοδοι κάποια στιγμή να εκπνεύσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο γιατί υπάρχουν και συμμετρίες σε τέτοιες συμφωνίες οι οποίες θα πρέπει κάποια στιγμή να τερματιστούν και όχι στο ειδικέ, ξέρω εγώ, για ακόμα 20 χρόνια να έχουμε αυτές τις ασύμμετρες εξελίξεις. Επιπλέον το Βιετνάμ παραμένει μια χώρα που το κράτος δικαίου ε, δεν είναι τόσο αναπτυγμένο ε, όσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα απέχει πόρο από αυτή. Έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα εδώ συμφωνίας όπου χρειαζόμαστε και προστασία των επενδύσεων και εξασφαλίσουμε ότι οι επενδυτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Βιετνάμ θα προστατεύονται ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι το σύστημα τους δεν είναι σαν το δικό μας της ελεύθερης δημοκρατίας και να έχουν κίνητρα οι επενδυτές να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο Βιετνάμ γνωρίζοντας ε, ότι θα προστατεύονται από την αυθαιρεσία της κυβέρνησης και από την πολιτική επιρροή ε, των αποφάσεων των δικαστηριών. Θα πρέπει να υπάρχει μια προστατευτική ε, ασφαλιστική δικλίδα για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Ε, ελπίζω να υπερψηφιστεί το ψήφισμά μας σήμερα. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόοδο των ε, διαπραγματεύσεων. Ήταν φιλόδοξος ο στόχος μας να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις εντός του έτους και θα ήμουν ευγνώμων αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους επόμενους μήνες ε, τηρήσει αυτή τη δέσμευση και ευχαριστώ και το Βέρνερ Λάγκε που είναι και παρόν σήμερα, το επικεφαλής της αντιπροσωπείας ΑΣΕΑΝ και όλη την αντιπροσωπεία και θα ευχόμουν στην αρχή της επόμενης θητείας να ολοκληρωθεί και να έρθει αίσιο πέρα αυτή η συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Ο κύριος Μπέντ Λάγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Μάλιστα, και εμείς είμαστε ακράδαντα πεπισμένοι ότι το εμπόριο, ε, η φόρος ε, ε, είναι κάτι που ενισχύει την αηφόρο ανάπτυξη και γι' αυτό υποστηρίζουμε και τις διαπραγματεύσεις με το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ είναι μια χώρα που μέσω του εμπορίου μπορεί να δημιουργήσει ευημερία για τους ανθρώπους, για το λαό του και οι 7 γύροι διαπραγματεύσεων ε, υπόσχονται πολλά, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι η ευημερία και η εφορία μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο εφόσον είναι δίκαιες οι συνθήκες και οι όροι. Και υπάρχουν τρεις τομείς εκεί που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Πρώτον, προστασία των ζώων και ο σεβασμός ε, των διεθνών κανόνων. Υπάρχει η σύμβαση ΣΑΙΤΕΣ για το παράνομο εμπόριο ε, σπανίων ειδών πανίδας. Το δεύτερο είναι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία και το τρίτον, το τρίτο πώς θα εξασφαλίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, οι προδιαγραφές για το περιβάλλον και οι κοινωνικές προδιαγραφές να τηρούνται. Ιδιαίτερα στη δράση των εταιριών στο Βιετνάμ. Δηλαδή να είναι πιο δεσμευτική όλοι αυτή η όρη και η αηφορία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρινάλντι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε εδώ τα συνήθη ε, που επικρίνουμε σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Και αυτό το βλέπουμε και στην περίπτωση του Βιετνάμ όπως και σε άλλες διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, θα ήθελα η συμφωνία να μην γίνει εις βάρος της πρόσβασης ε, σε γενώσιμα φάρμακα για τους Βιετναμέζους. Πρωτίστως όμως, και αυτό το λέμε με απόλυτη σαφήνεια προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας κανόνας για duty drawback και κανένας κανόνας εις βάρος των, ε, ε της καταγωγής. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε για το Βιετνάμ είναι ότι πρόκειται για δικτατορία. Δικτατορία ε, με όλα τις ε, τα κομφόρ, ε, καταπίεση μειονοτήτων, ε, οι βουδιστές αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ε, οι χριστιανοί που ζουν στις ορεινές περιοχές διώκονται και υπάρχει ένα κόμμα το οποίο αφήνει ελάχιστο περιθώριο ελευθερίας της έκφρασης στην κοινωνία των πολιτών. Υπάρχουν blog ιστολόγια τα οποία ε, διώκονται ή κλείνουν. Και θα θέλαμε να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το θέμα της ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, τι γίνεται με τους μηχανισμούς αξιολόγησης και ίσως και ανιστολής της συμφωνίας σε περίπτωση που τα όσα ζητάμε για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν γίνουν σεβαστά και επίσης το άνοιγμα των αγορών μας να μην είναι αυτός σκοπός για την αύξηση των υπαρικών συναλλαγών, αλλά να είναι πραγματικά ένας τρόπος προόδου του Βιετνάμ. Και η ε, συμφωνία ακριβώς για αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και πολύ πιο ευαίσθητη από συμφωνίες που κάναμε με άλλες χώρες ε, και μία ακόμα δικτατορία όπως για παράδειγμα τη Σιγκαπούρη. Και ελπίζω ότι το επόμενο ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι πιο απαιτητικό από εμά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζάραντελ. Ζάχραντελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Κύριε Επίτροπε. Είχα την τιμή να είμαι μόνιμος εισηγητής για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών στην Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου και ήταν τιμή για μένα για δύο λόγους. Ο ένας είναι το γεγονός ότι το Βιετνάμ είναι μια χώρα που ευημερεί και θα είναι πολύ καλός εμπορικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δεύτερος λόγος είναι συμβολικός. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι η κοινότητα των Βιετναμέζων στη χώρα μου, στην Τσεχική Δημοκρατία, είναι κατά αναλογία η μεγαλύτερη ε, κοινότητα Βιετναμέζων στις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως ήταν και αυτός ένας από τους λόγους που με τα χαράς ανέλαβα τα καθήκοντα του εισηγητή. Ο εισηγητής ε, διαπίστωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ε, προχωρέουν ε, και υπάρχει περιθώριο συνεννόησης ε, μεταξύ των δύο μερών σε αρκετά κεφάλαια και ελπίζω να είναι μια συμφωνία ε, προς όφελος όλων η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Νομίζω ότι εγκρίναμε ένα ισορροπημένο ψήφισμα το οποίο στόχο έχει να συνεισφέρει στην επιτυχία των διαπραγματεύσεων και Διευκρινίσαμε κάποιες προτεραιότητες όσον αφορά αυτές τις διαπραγματεύσεις και θα ήθελα να επισημάνω κάποιες από αυτές τις προτεραιότητες. Αυτό το οποίο θα θέλαμε είναι όλες οι διατάξεις οι οποίες είναι διαπραγμάτευση... σε αυτή τη Συμφωνία Ελευθέρων Συνολογών να είναι συμβατές με τις, ε, τα όσα προβλέπει ο ΠΟΕ, να υπάρχει πλήρη άρση των ε, περισσότερων δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών και θα θέλαμε να υπάρχει αμοιβαίο σεβασμό ω προ την δυνατότητα του να νομοθετούν, κυρίω στο θέμα των δημοσίων υπηρεσιών να ε, υπάρχουν κανόνες ανταγωνισμού ώστε να υπάρχουν θεμητοί όρια ανταγωνισμού μεταξύ των ε, βασικών παρόχων υπηρεσιών και μεγάλων επιχειρήσεων και να υπάρχουν και ε, διατάξεις για τη διαφάνεια και την επίλυση διαφορών ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Επίσης και οι δύο πλευρές θα πρέπει να δεσμευτούν για την εφαρμογή των πνευματικών δικαιωμάτων και θέματα υγεία και φυτοϊγείας και τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, και οι δύο πλευρά να σέβονται και ε, να συμμορφούνται με τα διεθνή πρότυπα στον τομέα των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικών συμφωνιών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο της, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και συζητητέ ε, για την επικοδομητική συνεργασία και ελπίζω να εγκριθεί από την Ολομέλεια το κείμενο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος ε, Μέρφυ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό το ψήφισμα ουσιαστικά είναι το ελεύθερο δικαίωμα για να κάνουν οι Ευρωπαίοι μεγάλες business για να προχωρήσουν ε, στην ταχεία ολοκλήρωση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών με το Βιετνάμ. Βεβαίως έχουμε τα συνήθη υποχρεωτικά, ε, την πρόσβαση στα φάρμακα, εταιρική ευθύνη, ε, δικαιώματα των ζώων, κοινωνικά, αλλά βασικά η αμοιβαία λέει άνοιξη των αγορών, απελευθέρωση, ιδιωτικοποίηση ε, και παραθέτω για να υπάρχει εγγυημένος ελεύθερος ανταγωνισμός. Καλή για ένα μηχανισμό διευθέτησης των διαφορών των επενδυτών για να μπορούν οι εταιρείε να την κυβέρνηση ε, όταν αυτό αντιβαίνει στα ε, κέρδη του. Η Occidental Petroleum με πετρελαϊκή των Ηνωμένων Πολιτειών ε, ζητάει 1,3 εκατομμύρια δολάρια κατά τη κυβέρνηση του Ισημερινού για εκμετάλλευση πετρελαίου στον Αμαζόνιο. Αυτά είναι καταπάτηση των δικαιωμάτων, παιδική εργασία και άλλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά δικαιώματα που παραβιάζουν. Ευχαριστώ. Κύριος Μπάστιαν Μπέλντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ είμαι. Αν δεν με βλέπετε από εκεί που είστε. Κύριε Πρόεδρε, το ψήφισμα που καλούμε θα σήμερα να ψηφίσουμε ε, ορίζει ε, ε, ένα διμερή διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούνται σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας ζητήσω την προσοχή σας για την δινή θέση στην οποία βρίσκονται οι χριστιανοί στο Βιετνάμ. Αναφέρθηκε και προηγουμένως. Πρόσφατα μία ΜΚΟ Open Doors έφερε ένα κατάλογο με χριστιανούς που διώκονται στο Βιετνάμ. Πέρσι ήταν στη 40η θέση και φέτος στη 18η το Βιετνάμ. Παραβιάζει τα δικαιώματα ε, των χριστιανών στην ε, επαρχία την ορεινή. Ε, υπάρχουν περιορισμοί στις θρησκευτικέ ελευθερίες με βάση ένα νέο νόμο. Τα θρησκευτικά ιδρύματα θα πρέπει να ζητούν την άδεια για να διοργανώσουν τη λατρεία και τις λειτουργίες τους. Και αυτό ε, πραγματικά είναι εξωφρενικό. Διώκονται οι, οι καθολικοί από τις ίδιες τους συστίες. Τους στέλνουν την αστυνομία, τις διοκτικές αρχές, ακόμα και το στρατό. Ε, και καταστρέφουν ε, τα σπίτια τους, τα ισοπεδώνουν κυριολεκτικά. Παρακαλώ να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανεξιθρησία και θα πρέπει να το θέσουμε υπόψη των Βιετναμέζων το συνομότερο. Η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να είναι κενό γράμμα, αλλά να είναι ουσιαστικό στοιχείο της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Herr Ο κύριος Φρανκ Προύστ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Τα τελευταία χρόνια Είχαμε αποτυχία της, ε, ε, μεγάλη επιτυχία της Ασίας ε, ως οικονομία παγκόσμια οικονομία, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Οι ασιατικές χώρες έχουν ποσοστά ανάπτυξης της τάξης του 5 ή του 6% και πολλές φορές και διψήφια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραμείνει αδρανή ενώπιον αυτών. Αναφερόμαστε σε αναδυόμενε χώρες συνεχώς, ε, οι οποίες, ε, χώρες οι οποίες μετατράπηκαν τώρα σε ισχυρές οικονομίες και θα πρέπει ε, να μπορούμε να δούμε και εμεί τι θα κάνουμε. Πολλές φορές από αφέλεια ή από υπεροψία αγνοήσαμε αυτές τις απαιτήσει και τώρα ήγηκε η απο υπεροψια αγνοησαμε αυτέ τι απαιτησει και τωρα και η ωρα να τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Η Εκείνα είχε ανάπτυξη της τάξης του 5% και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ίδιο ισχύει και για το Βιετνάμ. Πρόκειται για μια χώρα με την οποία δεν μπορούμε να μην έχουμε ε, οικονομικές συναλλαγές. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν οι διαπραγματεύσεις με το ε, Βιετνάμ με στόχο Συμφωνία Ελευθέρωσης Αναγών και ε, θα πρέπει αυτές να οδηγήσουν σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα για τις δύο πλευρές. Ω ευρωπαϊκή χώρα εμείς θα πρέπει να διατηρήσουμε τα συμφέροντα των ε, σημαντικών μας επιχειρήσεων και των πιο σημαντικών τομέων με στόχο το άνοιγμα αυτών των αγορών και επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε η συμφωνία αυτή να είναι προς όφελος κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Βιετνάμ εισάγει ε, ευρωπαϊκά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες σε θέματα τεχνολογικά. Και αυτό είναι το μόνο ανταγωνιστικό προλέκτημα που έχει η Ευρώπη σε σχέση με τους υπολείπους. Είμαι πεπισμένος ότι χάρη σε αυτή την ε, τεχνολογική τεχνογνωσία θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεν πρέπει να σταματήσουμε ενώπιον αυτής ε, της προόδου της Ασίας. Θα πρέπει μαζί να συνεργαστούμε για να έχουμε μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη διεθνώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω αυτές τις διαπραγματεύσεις αλλά πιστεύω όπως και οι συνάδελφοι το θέμα θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από την απλή διάνοιξη των αγορών. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε καταρχάς ότι οποιαδήποτε συμφωνία προάγει την ε, δίκαιη ανάπτυξη ε, στο Βιετνάμ. Υπάρχει το θέμα της αρπαγής γεών που είναι τεράστιο θέμα στο Βιετνάμ και εγώ δεν θέλω μια τέτοια συμφωνία να διευκολύνει περαιτέρω αρπαγή γεών από ευρωπαϊκές ή άλλες εταιρείες. Δεύτερον, σε κάθε τέτοια ε, συμφωνία θα πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό κεφάλαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη. Για μας είναι κόκκινη γραμμή για την πολιτική μου ομάδα. Για την ευημερία των ζώων πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνεται σε οποιαδήποτε συμφωνία με το Βιετνάμ. Η κατάσταση της πανίδας εκεί ε, είναι πραγματικά εξωφρενική και των ζώων γενικότερα. Και Έχουμε ήδη ένα προηγούμενο και ένα υπόδειγμα που είναι η συμφωνία με την Κορέα. Εφόσον συμφωνήσαμε με την Κορέα μπορούμε να τα βρούμε και με το Βιετνάμ. Και αυτό είναι ένα προπομπό γενικότερα για μια περιφερειακή συμφωνία και θα πρέπει το συντομότερο να επιτευχθεί συμφωνία με όλε τι χώρε ε, ΑΣΕΑΝ, τη Νοτιοανατολική Ασία. Ευχαριστώ, κύριο Μπιέλαν. Κύριε Πρόεδρε, Ένα σύστημα ελευθέρου εμπορίου αντανακλά την ανάγκη να υπάρχει ελεύθερο εμπόριο σε διεθνέ πλαίσιο και αυτό φυσικά είναι προ όφελο των πολιτών. Το Βιετνάμ είναι μια πολύ δυναμική οικονομία, ε, μία από τι χώρε που συμμετέχει στην ΑΣΕΑΝ και ε, ε, φτάνει σε 8% ανάπτυξη του ΑΕΠ ετησίω. Και ελπίζω λοιπόν να μπορέσει να ολοκληρωθεί η συμφωνία μέχρι το τέλο του έτου ώστε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μα με τον εταίρο αυτό. Μα ενδιαφέρει ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται σε ελεύθερο και θεμητό ανταγωνισμό και η δασμολογική και δι, μη δασμολογική φραγμή προς το εμπόριο θα πρέπει να αρθούν. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ε, το Βιετνάμ είναι μια χώρα στην οποία εξακολουθούν να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ θα πρέπει να μεταφράζεται και σε ενίσχυση αυτών των δικαιωμάτων. Κύριο κύριος Λάγκεν, πρόεδρος της αντιπροσωπεία με τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι έχει δίκιο ο κύριος Αλμούνια. Ε, είναι success story το Βιετνάμ από πλευρά οικονομία. Καλύτερα ε, μια συμφωνία με όλες τις χώρες ΑΣΕΑΝ έχει δίκιο και ο Ντέιβιτ Μάρτιν. Γιατί είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές ε, από χώρα σε χώρα όμως αυτή τη στιγμή για να έχουμε συνολική συμφωνία. Με πέντε χώρες κάνουμε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και μετά με 7 από τις δέκα συνολικά έχουμε συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας. Τα ζητήματα ε, όλα περιλαμβάνονται στην έκθεση του συναδέλφου Ζάχραντιλ. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα και νομίζω ότι οι καλέ οικονομικέ σχέσει και η οικονομική ελευθερία θα πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι με την ελευθερία τη σκέψη, τη άποψη και τη θρησκεία. Και τα γνωρίζουν αυτά οι εταίροι στο Βιετνάμ. Την τελευταία φορά που πήγα εκεί, το φθινόπωρο του 2013, το συζήτησα αυτό με όλου του διαπραγματευόμενου και του εταίρου μα εντατικότατα και εξεπλάγει ε, από ε, την έλλειψη θάρρου από το Κομμουνιστικό Κόμμα για να γίνουν μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Υπάρχει μια ιστορία και λυπάμαι που το τελευταίο συνέδριο τους δεν επέτρεψε αυτό το άνοιγμα. 35 ε, εκατομμύρια πρόσβαση στο ίντερνετ έχουν στο Βιετνάμ ε, και παρόλο αυτά αν πούν κάτι οι bloggers που αντιτίθεται στο καθεστώς είτε τους κόβουν το διαδίκτυο είτε τους συλλαμβάνουν. Πού είναι οι ελευθερίες, πού είναι η σύγχρονη χώρα. Και είναι σωστό το Κοινοβούλιο να καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να την πιέζει να κάνει συνολικά διαπραγματεύσεις. Θα χαιρόμουν να ολοκληρωθούν φέτος αυτές, οπωσδήποτε, αλλά το επόμενο βήμα και το επόμενο στάδιο που έχουμε σε πολλές συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών θα πρέπει επίσης να επιταχυνθεί, που είναι η κύρωση πλέον από τα 28 κράτη-μέλη. Τι νόημα έχει να εργαζόμαστε εμεί σκληρά και γρήγορα και τα κράτη-μέλη να χρονοτριβούν στην κύρωση. Γι' αυτό χαίρομαι για τι διαπραγματεύσει και εύχομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπαντία Ικουτσέτ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Ευθύ εξ αρχή αυτή τη συμφωνία ελευθέρου συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Βιετνάμ το 2012 έγιναν πολύ σημαντικά βέματα για να μπορέσει να καθοριστεί η συμφωνία και να ολοκληρωθεί. Χαίρομαι για την πρόοδο που έχει επιτύχει το Βιετνάμ σε θέματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών δικαιωμάτων και ελπίζω αυτή η συμφωνία να αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα για τη διεύρυνση αυτών των δικαιωμάτων. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και ένα κεφάλαιο για βιώσιμη ανάπτυξη με δεσμευτικού όρου ώστε να αποτελέσει και ακρογωνιαίο λίθο ε, για το Βιετνάμ όπως είναι και για την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, τα αμοιβαία συμφέροντα και οι διαχωριστικές γραμμές ε, κατέρωθεν δεν θα πρέπει να αποτελέσουν ανάχωμα στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, διότι η συμφωνία αυτή σίγουρα θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική ευκαιρία και για τις δύο πλευρές σε τομείς όπως είναι οι εμπορικές ροές και άμεσες ξένες επενδύσεις και επίσης θα πρέπει να επενδύσει επενδύσουμε και στην ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής ΑΣΕΑΝ και ελπίζω να υπάρχουν και κάποιες μελλοντικές συμφωνίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριο Σκέλη. Ε, ε, ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και άλλοι μιλητές, καλωσορίζω αυτήν την διαπραγματεύσεις ελευθέρων συναλλαγών, εμπορικών συναλλαγών με το Βιετνάμ. Ολοκληρώσαμε διάφορες συμφωνίες με τον Καναδά, τη Νότια Κορέα και άλλες ε, και αξίζει τον κόπο να έχουμε μια τέτοια συμφωνία και με το Βιετνάμ, το οποίο αξίζει μεγάλους επένους για την πρόοδο που έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Πριν από κάποια χρόνια δεν ακουγόταν τίποτα για το Βιετνάμ εκτός και από, από ε, ε, πόλεμο νεκρούς και τέτοια. Τεράστια πρόοδος λοιπόν. Ε, συμφωνία ε, για 23,8 δις ε, ε, Έχουμε δηλαδή 8 εκατομμύρια στις εξα... δισεκατομμύρια στις και ε, τα αντίστοιχα για τις ε, εξαγωγές. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν από αυτή την άποψη να δούμε να αφήσουμε τις επιχειρήσεις μας να εξάγουν περισσότερο προς το Βιετνάμ. Και επιπλέον δίνουμε ε, την ευκαιρία στους δικούς μας ε, ανθρώπους να ξεφύγουν από την κρίση η οποία μας ταλανίζει τόσα χρόνια ταυτόχρονα. Όπως είπαν και άλλοι ομιλητές, είναι πολύ σημαντικό να σέβεται το Βιετνάμ τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία, την ελευθερία έκφρασης και την ελευθεροτυπία και πιστεύω πως θα μπορέσουμε όντως να προχωρήσουμε και σε αυτούς τους τομείς γιατί στο τέλος αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτή και ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις πριν το τέλος του έτους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Δεν έχουν ζητήσει συνάδελφοι το λόγο στη διαδικασία Catch οπότε θα παρακαλέσω τον Επίτροπο κύριο Αλμούνια να κλείσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ επίσης όλους τους βουλευτές ε, που μιλήσατε ε, στη συζήτηση αυτή. Οι περισσότερες παρεμβάσεις συμπίπτουν με τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πρόκειται για μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών η οποία ή δυνατόν θα πρέπει να ολοκληρωθεί ε, εντός του έτους και να είναι θετική και θα είναι θετική για πολλούς λόγους και αμοιβαίως επωφελής. Ε, θα ήθελα να μοιραστώ ε, μαζί σας μερικά σχόλια και ανησυχίες που ακούστηκαν στις παρεμβάσεις σας. Πρώτον, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ε, οικονομικοί και εμπορικοί μας εταίροι να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα αντιμετωπίζουμε στο θεσμικό μας διάλογο, εταιρική σχέση και συνεργασία στη συμφωνία μας με το Βιετνάμ και θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων που μπορεί να κινδυνεύουν στη χώρα αυτή. Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, ε, καλύπτονται αυτά τα ζητήματα στο κεφάλαιο αϊφόρου ε, ε, ανάπτυξης, συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, το κείμενο όπως έχει τώρα και όπως το διαπραγματευόμαστε και οι διαπραγματευτές μας συμφώνησαν και μάλιστα έτσι με στεναρή γλώσσα για θέματα που έχουν να κάνουν με το Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας και τις αντίστοιχες διατάξεις που ε, διέπουν την προστασία της εργασίας. Και κάποια άλλα στοιχεία που αναφέρατε, η προστασία των ζώων, το Βιετνάμ συμφώνησε να συμπεριλάβει τα ζητήματα αυτά στη συμφωνία Ε, προτιμά ε, να τα συμπεριλαμβάνει αυτά στο κεφάλαιο εμπόριο και αηφόρος ανάπτυξη. Εμείς θέλουμε να μπει στο κεφάλαιο που αναφέρεται στα ε, υγειονομικά και φυτοϊγειονομικά μέτρα. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις, σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και ελπίζω στο επόμενο κοινοβούλιο, τους επόμενους μήνες να είμαστε σε θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας ενημερώσει για την επιτυχή έκβαση και ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Για να κλείσει λοιπόν η συζήτηση, πρέπει να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι η αρμόδια Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ε, κατέθεσε ψήφισμα. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Η δε ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 12 το μεσημέρι. Και περνούμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης. Σύντομη παρουσίαση της ακόλουθης έκθεσης. Είναι η έκθεση του κυρίου Πέτερλε με θέμα της διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής.